και τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Ε, θα ενημερώνουμε συνεχώς το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Τεχόχτ. Έχω λάβει δύο ψηφίσματα. Ε, το ένα είναι από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και το άλλο από την ομάδα των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη σας λέγω ότι δεν έχει ζητηθεί να ε, ψηφιστούν εκθέσεις που πρόκειται να διαδοθούν μέχρι τις 5.30 και θεωρούνται εγκεκριμένες.